αυτές οι αποφάσεις. Διάφορες επιτροπές έχουν αποφάσει να αρχίσουν ε, διοργανικές διαπραγματεύσεις με το άρθρο 69 γάμου παραγράφος 1 του κανονισμού και ε, υπάρχουν ε, ε, σχετικά πρακτικά στην ε, ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Και δυνάμει του άρθρο 69 γάμου παραγράφος 2 τα μέλη κάποιες πολιτικές ομάδες με αριθμό που προβλέπετε ε, πρόκειται να ζητήσουν εγγράφος αύριο να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για τις οποίες να γίνει ψηφοφορία. Επίσης, ε, θα αρχίσουν